All right, everybody, welcome. Καλώς ορίσατε, απαντές. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Καλώς ορίσατε, απαντές. Παρακαλώ, μ' αρέσει να χτυπάω το σφυράκι. Πολύ γέλιο. Καλώς ορίσατε όλοι. Το μέλλον της βιομηχανίας μεταποίησης ε, στην Ευρώπη είναι ένα πιλωτικό έργο που αρχικά είχε προταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, από τον Μεδρίλ, πρώην συντονιστή της Ήτρε, είχε συμφωνηθεί για το δημοσιονομικό έτος 2014 και 2015 ε, ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Eurofound, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Βελτίωσης των Συνθήκων Εργασίας και Διαβίωσης. Οι συντονιστές ε, και των δύο επιτροπών, Ήτρε και Έμπλα, ε, βρίσκονται εδώ για να ακούσουν τα ευρήματα αυτού του κοινού έργου για την ανταλλαγή αυτή δείχνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα επειδή η Κομισιόν πρόσφατα δημοσίευσε μια ανακοίνωση για μια ανανεωμένη βιομηχανική πολιτική. Η Επίτροπος Βιενκόφσκα παρουσίασε τα κύρια χαρακτηριστικά στη συνάντηση της Ήτρε της Δευτέρας Οκτωβρίου. Η Ήτρε αποφάσισε να δώσει συνέχεια σε αυτή την ανακοίνωση με μια προφορική ερώτηση προς ε, την Κομισιόν. Χαιρόμαστε λοιπόν που θα γίνει αυτή η κοινή συνεδρίαση σήμερα και να δώσω το λόγο σε εσάς κυρία Ολσκό για μια εισαγωγή και για να προεδρεύσετε αυτή την παρουσίαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και εγώ φυσικά ήθελα να καλωσορίσω όλους τους συμμετέχοντες, ειδικότερα τους συναδέλφους και εμπειρογνώμονες της Eurofound, που θα μοιραστούν μαζί μας τα πρώτα ευρήματα αυτού του πιλωτικού έργου. Χαιρόμαστε που συνδιοργανώνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων φυσικά με την Επιτροπή Ήτρε. Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όπου έγινε μια πρώτη εστίαση στον τομέα των υπηρεσιών την τελευταία δεκαετία, παρατηρήσαμε να επανακτάξει η μεταποίηση ως δημιουργός θέσεων εργασίας και ανάπτυξης της οικονομίας μας. Για το σκοπό αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε την πρωτοβουλία αυτού του πιλωτικού έργου που ανέφερε ο συναδελφό μου το μέλλον τη βιομηχανία μεταπίση στην Ευρώπη, που ξεκινάει από το 2015 μέχρι το 2019 και που ανατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Βελτίωση των Συνθήκων Εργασία και Διαβίωση, το Eurofund εν συντομία. Η μεταποίηση, η έρευνα και η ανάπτυξη εξελίσσονται παράλληλα. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό και φυσικά γνωρίζουμε ότι είναι ζωτική σημασία για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πρέπει οπωσδήποτε να μην ξεχνάμε ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα των εξαγωγών της Ευρώπης σήμερα είναι μεταποιημένα αγαθά. Το λέω αυτό διότι είναι ότι το ξεχνάμε η ταχεία πρόοδος και η τεράστια κλίμακα τεχνολογικής καινοτομίας σήμερα θα επιφέρουν τεράστιες αλλαγές στον τομέα της μεταποίησης. Οι συνέπειες ε, δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν. Ορισμένοι παρατηρητές ε, αναφέρονται μάλιστα σε νέα βιομηχανική επανάσταση. Σε έναν κόσμο όλο ένα και πιο παγκοσμιοποιημένο, όπου οι παράγοντες ε, παραγωγής, οι συντελεστές παραγωγής ε, είναι ε, μοιρασμένοι σε όλο τον κόσμο. Είναι σημαντικό η Ευρώπη να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της και να διασφαλίσει την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας για τους Ευρωπαίους. Κάτι πολύ ανησυχητικό αυτών των νέων εξελίξεων είναι ότι η παραγωγή, η μεταποίηση προβλέπεται να απαιτεί λιγότερα εργατικά χέρια αυτή η απώλεια θέσεων εργασία ε, στον τομέα τη μεταποίηση θα πρέπει να εξισορροπηθεί, να αντισταθμιστεί με δημιουργία θέσεων εργασία αλλού, σε άλλου τομεί παραγωγή. Όπω έγινε τι τελευταίε δεκαετίε ε, του τελευταίου αιώνα, όταν ο τομέα μεταποίηση μα ε, υπέστη τι πρώτε συνέπειε τη παγκοσμιοποίηση ζητήματα. Όλα αυτά πολύ ενδιαφέροντα για την Επιτροπή Απασχόλησης και για τις εργασίες αυτής της ομάδας είναι το πώς αυτές οι νέες ε, εξελίξεις επηρεάζουν τις θέσεις εργασίας, ε, τα εισοδήματα, την κοινωνική ασφάλιση, τα εργασιακέ εργασιακές συμβάσεις, ε, τα μοντέλα εργασίας, τις δεξιότητες και την κατάρτιση. Πρέπει όμως επίσης να διασφαλίσουμε και το ότι δεν θα αφήσουμε πίσω τους πιο ευάλωτους πολίτες, ε, ότι οι κοινωνίες μας ε, θα έχουν τη συμμετοχή όλων. Ε, πολλοί κερδίζουν στην αγορά εργασίας, αλλά κάποιοι υπάρχει κίνδυνος να βρεθούν στη θέση του χαμένου, των χαμένων. Και σήμερα είναι υποχρέωσή μας να προσπαθήσουμε να τους κρατήσουμε όλους μαζί, θα εστιαστούμε σήμερα λοιπόν στο έργο του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι ύψη τη σημασία και αναμένω να ακούσω την παρουσίαση και την ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη. Ευχαριστώ. Uh, λοιπόν, θα δώσω τώρα το λόγο στην Eurofound και στην επικεφαλή της έρευνας τον κύριο Στόρι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την πολύ καλή εισαγωγή σε ό,τι αφορά το θέμα του μέλλοντος της μεταποίησης. Βεβαίως ε, και πρέπει να το εξετάσουμε το μέλλον αυτό από πλευρά ε, βιομηχανικής πολιτικής, ε, πολιτικής απασχόλησης, οικονομικής πολιτικής της Ένωσης διότι υπάρχουν οι τεχνολογικές εξελίξεις μεταξύ άλλων ε, οι οποίες λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή. Εγκρίθηκε το πιλωτικό πρόγραμμα το 2013 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ουσιαστικά πρόκειται για προγράμματα έρευνας στο έγγραφο εκείνο του Κοινοβουλίου. αναφέρω εδώ μια σειρά από παραπομπέ, Συμφωνία με την Κοινική Διεύθυνση GROW ε, υπογράφηκε τον, 15 Απριλίου του 2015 με ολοκληρώση τον Απρίλιο του 2019 Είχαμε συζητήσει με την DG Grow που συνεισέφερε σημαντικά σε ό,τι αφορά του διάφορου τομεί έρευνα που είχαν προταθεί και έχουμε πλέον ένα reshoring monitor το οποίο θα δίνει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητε στον τομέα της μεταποίησης και της καινοτομίας, στον τομέα αυτών. Ιδιαίτερα στα πλαίσια της νέας πολιτικής συνοχής ε, εξετάζεται το θέμα της δυνατότητας, δυνατοτήτων που υπάρχουν σε επίπεδο μηχανικής πολιτικής και δεν αναφερθώ σχετικά. Πολύ πολύ χρήσιμο για μας αυτό το, ε, αυτή η ομάδα, η διαπηρεσιακή, συναντιέται δύο φορές το χρόνο. Η υπηρεσιακή ομάδα λοιπόν ε, από την Επιτροπή ε, από διάφορε διάφορα τη Επιτροπή και από του κοινωνικού εταίρου μεταξύ άλλων. Έχουμε προετοιμάσει και μια σειρά ακόμα διαφάνειε για το European Resource Monitor. Αναφέρθηκα προηγουμένω. Επλέον θέλω να πω κάτι. Επειδή έχω μόνο 10 λεπτά, θα πρέπει να είμαι εξαιρετικά έτσι, σφιχτό στην παρουσίασή μου. Ένα μεγάλο μέρο ένα μεγάλο υπο-project ε, σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα είναι τα ποσοτικά σενάρια για το μέλλον της ε, μεταποίησης στην Ευρώπη. Από αυτού εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο βεβαίως ε, να οδηγηθούμε σε συγκεκριμένα σενάρια που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν με οικονομικό τρόπο ε, για ένα τόσο περίπλοκο και μακροοικονομικό μοντέλο. Έχω όμως κάποια πρώτα αποτελέσματα τα οποία θα μπορούσα να σας ε, αναφέρω σε ό,τι αφορά την απασχόληση στην Ευρώπη, ένα σενάριο παραδείγματο χάρη στον τομέα τη μεταποίηση ε, πιο συγκεκριμένα, ε, με τον πλήρη σεβασμό βεβαίω πάντα και των, ε, Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, ε, τα αποτελέσματα ε, μας δείχνουν εδώ ότι έχουμε ένα συνολικό μοντέλο, ε, σφαιρικό μοντέλο, εξετάσουμε και γίνεται και αλλού στον κόσμο δηλαδή, και τα αποτελέσματα για την Ευρώπη, εν περιπτώσει, είναι εξαιρετικά. Ε, αυτό βεβαίως είναι το ελκυστικό σενάριο ε, για την Ευρώπη με την Συμφωνία των Παρισίων. Χρειάζεται βεβαίω σημαντική ε, επένδυση δημόσια στην αρχή με τον ε, πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που μια κινησιανής ας πούμε πολιτικής ιδιαίτερα στον τομέα της μεταποίησης ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν σύμφωνα με αυτό το σενάριο με βάση βεβαίω τι επενδύσει που θα λάβουν χώρα, τι δημόσιε επενδύσει για να γίνουν σεβαστή η Συμφωνία των Παρισίων, σημαντική αύξηση τη απασχόληση στη Γερμανία, αλλά, αλλά ε, έχουμε επίση σημαντικέ αυξήσει στην απασχόληση και στη Γαλλία, την Ισπανία, το οποίο μπορεί να εκπλήξει προ τι αλλά δεν είναι και τόσο περίεργο. Γνωρίζω ότι δεν έχω πολύ χρόνο. Τώρα για το monitor αυτό, δηλαδή αυτό, αυτό το σύστημα ε, συλλογής δεδομένων από διάφορους, ε, ε, διάφορες πηγές, οργανώσεις, κλαδικές, περιοδικά εξειδικευμένα. Προσπαθούμε λοιπόν να συλλέξουμε στοιχεία σε ό,τι αφορά την επιστροφή των εργαζομένων στον τομέα αυτών στην Ευρώπη. Δυστυχώς ε, τα βασικά ευρήματα που έχουμε είναι ότι είναι μικρές επιπτώσεις για την απασχόληση αυτής, αυτού του εγχειρήματο. Από τι 150 υποθέσεις που εξετάσαμε, μόλις 21 εξ αυτών ε, δημιούργησαν πάνω από 100 θέσεις εργασίας. Ε, δεν είναι λοιπόν μια σημαντική πηγή απασχόλησης, αύξηση της απασχόλησης στην τομέα τη μεταπίσης για την ώρα τουλάχιστον. Είναι βεβαίω μια πλούσια πηγή πληροφοριών. Ε, ποιε επιχειρήσει ε, επιστρέφουν, ποιε λειτουργίε τη επιχείρηση επέστρεψαν πιο συγκεκριμένα στην Ευρώπη. Επίσης ε, κάποια στοιχεία για τις προσπάθειες που γίνονται στα διάφορα κράτη-μέλη. Πριν απο τρία-τέσσερα χρόνια ήταν ε, δημοφιλές το θέμα αυτό. Είχαν γίνει και μια, πρωτο, σειρά πρωτοβουλίε και στη Γαλλία, στην Ιταλία και στον Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές οι πρωτοβουλίες ε, όμως ε, δεν είχαν συνέχεια, δεν είχαν τους απαραίτητους πόρους, ε, δεν δόθηκε όπως μια στεναρή συνέχεια και σε ό,τι αφορά τι δραστηριότητε λοιπόν τη επιστροφή τη απασχόληση, ε, που συμβαίνουν αλλού στον κόσμο, ε, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού Παραδείγματο χάρη, ε, θα πρέπει και εμεί να κάνουμε μια προσπάθεια να ενισχύσουμε αυτή, την, αυτά τα project. Εντάξει, όχι να πάμε απαραίτητα η Ευρώπη πρώτα, αλλά θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο και εμεί το θέμα αυτό. Να δώσω το λόγο στη συνάδελφο. Ένα άλλο project ερευνών που καλύπτουμε εδώ έχει να κάνει με την πολιτική προοπτική, την περιφερειακή βιομηχανική πολιτική. Και εδώ εξετάσαμε πιο συγκεκριμένα ποιε είναι οι δυνατότητε που υπάρχουν στο περιφερειακό επίπεδο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων ε, τη πολιτική αυτή. Εδώ αναλύουμε εννέα διαφορετικούς τομείς σε όλη την Ευρώπη και προσπαθούμε να διερευνήσουμε του προσανατολισμού της ε, περιφερειακής βιομηχανικής πολιτικής, ποιοι είναι οι φορείς που συμμετέχουν, ποιες είναι οι διαδικασίες σχεδιασμού της εφαρμογής ε, της βιομηχανικής πολιτικής, τι μπορεί να προσδιοριστεί ως καλή πρακτική προκειμένου να επιτυγχάνονται ε, πραγματικά αποτελέσματα ε, μέσω αυτών των ενδιαφερουσών πρωτοβουλειών. Αυτό που βρίσκουμε λοιπόν είναι ότι σε περιφερειακό επίπεδο δεν υπάρχουν έγγραφα τα οποία να ε, ασχολούνται συγκεκριμένα με την περιφερειακή βιομηχανική πολιτική. Κυρίως ο όρος που χρησιμοποιείται είναι περιφερειακή ανάπτυξη. Ε, Παρ' όλα αυτά είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπάρχουν διάφοροι τομείς πολιτικής που καλύπτονται από, την, ε, από αυτόν τον όρο ομπρέλα. Για εσάς ε, αυτό που σας ενδιαφέρει πιο πολύ είναι η απασχόληση βεβαίως. Ε, αυτός ο τομέας όμως φαίνεται ότι ε, έμεσα μόνο επηρεάζεται από την περιφερειακή ανάπτυξη. Παρ' όλα αυτά υπάρχει γνώση όσον αφορά τις δεξιότητες αλλά και τις, τους προσανατολισμούς της μελλοντικής χάραξης της πολιτικής όσον αφορά τη βιομηχανία μεταποίησης. Τι βλέπουμε λοιπόν όσον αφορά τις ικανότητες ε, τις βιομηχανικές. Αυτές επηρεάζονται αφενός από, την, από τις θεσμικές δομές, τη διακυβέρνηση, τις, τους ανθρώπινους πόρους βεβαίως που καλούνται, ε, των θεσμών που καλούνται να διαχειριστούν αυτές τις διαδικασίες. Υπάρχει όμως εμπειρογνωμοσύνη και γνώση τόσο όσον αφορά την, ε, το σχεδιασμό αλλά όσο, τόσο όσο, και όσον αφορά την ανάλυση και την αξιολόγηση, την παρακολούθηση των πολιτικών. Υπάρχουν ε, Πάντω ε, σε πολλές περιφέρειες προβλήματα όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση και όποτε γίνεται παρακολούθηση και αξιολόγηση γίνεται με αποσπασματικά μέτρα και όχι ε, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής ή πολιτικής. Κάτι το οποίο βεβαίως ε, ε, επιστρέφει ε, στην χάραξη πολιτικής με τη μορφή προβλημάτων στο σχεδιασμό. Όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές υπάρχουν διάφορα στοιχεία όσον αφορά τη διακυβέρνηση πολιτικής, το μείγμα που ακολουθείτε, το σχεδιασμό της πολιτικής και μπορείτε να βρείτε πολλά στοιχεία όσον αφορά τις, ε, την, τα στοιχεία, πολλά στοιχεία όσον αφορά την πολιτική αυτή στην έκθεση που θα εκδώσουμε πολύ σύντομα Υπάρχουν πάντως πολλές διαφορές μεταξύ των περιφερειών ε, και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό πάντοτε να έχει κανείς κατά νου ε, το ευρύτερο πλαίσιο μιας πολιτικής εντός του οποίου ε, εφαρμόζεται μια βιομηχανική περιφερειακή πολιτική και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να μεταφέρει ένα προς ένα μια βέλτιστη πρακτική από τη μία περιφέρεια σε μια άλλη. Ε, πολλέ φορέ φορές ε, μας λένε ότι είναι λίγο επιστημονική φαντασία αυτό που κάνουμε. Πολλέ φορές έχουμε ε, νέα στοιχεία, βιοτεχνολογία, το ίντερνετ των πραγμάτων, ηλεκτρικά οχήματα. Ε, όλα αυτά είναι διαδικασίες οι οποίες θεωρούμε ότι βρίσκονται στο επίκεντρο αλλά και στην, στην πρώτη γραμμή ε, των εξελίξεων στον τομέα της τεχνολογίας. Ε, υπάρχουν εξελίξεις στη ρομποτική που επηρεάζουν όλους το τομείς. Ε, βεβαίως τα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και τα πρόσθετα είναι πιο, εξειδικευμένοι τομείς οι οποίοι δεν έχουν άμεσες επιπτώσεις σε όλους τους άλλους τομείς της οικονομίας. Αποτελέσματα των, της διαδικασίας παραγωγής. Εδώ βλέπετε μια επισκόπηση. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια συγκέντρωση των ψηφιακών πληροφοριών στην παραγωγή παραγωγής. Ε, χρησιμοποιούνται όλο ένα και περισσότερο ψηφιακές διεργασίες, διαδικασίες, κάτι που έχει πολύ συγκεκριμένες επιπτώσεις και στο εργατικό δυναμικό. Η General Electric, για παράδειγμα, ε, έχει ξεκινήσει ε, πλέον ε, ε, μαθήματα εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού της για την ψηφιοποίηση. Ακριβώς για να δρέψει τους καρπούς αυτής της διαδικασίας, αυτού του φαινομένου. Το μέλλον της μεταποίησης βεβαίως δεν αφορά μόνο την ε, δημιουργία ενός μιας μαύρης Ford. Αντιθέτως ε, θα περιλαμβάνει βεβαίως και τα προσαρμοσμένα ε, προϊόντα στις ανάγκες των εκάστοτε καταναλωτών σε μαζική κλίμακα όμως. Αυτό σημαίνει ότι ολοένα και περισσότερο θολώνουν οι γραμμές, τα όρια ανάμεσα στη μεταποίηση και τις υπηρεσίες. Είναι ένα φαινόμενο ευρύτερο που επιφέρει η ψηφιοποίηση. Και αφορά ολόκληρη την ε, ζωή, τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος όταν πια βρίσκεται στα χέρια του καταναλωτή. Πολύ σημαντικό στοιχείο επίσης είναι η αυξημένη αποδοτικότητα των πόρων. Ε, χρήση ενέργειας, ε, αξιοποίηση αποβλήτων, όλα αυτά είναι φορείς που συμβάλλουν στη διαδικασία που περιγράφουμε ε, υπάρχουν και πολλές συμπράξεις, συνέργειες ε, μεταξύ διαφόρων κλάδων. Να ολοκληρώσω λέγοντας ε, ορισμένα στοιχεία που αφορούν την απασχόληση. Δυστυχώς ε, θα υπάρξει δομική μείωση ε, στην ενωσιακή μεταποίηση. Οι θέσεις απασχόλησης στη βιομηχανία μεταποίησης θα συνεχίσουν να μειώνονται. Ωστόσο, αυτό μας επιτρέπει σε μεγάλο βαθμό να διεξάγουμε αυτές τις διαδικασίες μεταποίησης στην Ευρώπη, κάτι που σημαίνει ότι ενδέχεται να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας σε άλλους τομείς της οικονομίας. Υπάρχει μια επαγγελματική αναβάθμιση. Φαίνεται ότι όλο ένα και περισσότερο χρειαζόμαστε περισσότερους μηχανικούς, περισσότερους μάνατζερ, λιγότερους εργάτες, χειρόνακτες. Αναμένουμε να υπάρξει μια ε, ορισμένη επαναγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι πολύ ε, σημαντικά τα ωφέλη όσον αφορά την απασχόληση. Ε, ανάλυση δεδομένων, ασφάλεια δικτύων, όλα, αυτά, όλα αυτοί είναι τομείς οι οποίοι θα δουν μια αύξηση στην απασχόληση. Συνθήκες εργασίας τώρα θα μειωθεί η βαριά ε, μορφή ε, της εργασίας, της ανθρώπινης εργασίας, θα μειωθούν οι κίνδυνοι οι επαγγελματικοί στην εργασία. Ωστόσο, ε, τα δεδομένα μας δείχνουν ότι θα συνεχίσει να, υπάρξει, να υπάρχει ε, θέμα και πρόβλημα ε, αυτή τη φορά στο νέο κύκλο, δηλαδή στη νέα φάση ανάπτυξης, ε, στους εργαζόμενους που ασχολούνται με τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων. Ρομπότ παρίες. Έχουμε δει πολύ, πολλά τέτοια φαινόμενα σε ταινίε τα τελευταία χρόνια. υπάρχουν κίνδυνοι, πρέπει να επαγρυπνούμε. Επίσης υπάρχουν σενάρια βάσει των οποίων ο διαχειριστής ή ο διευθυντής μιας υπηρεσίας δεν είναι αλλά αλγόριθμος και καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να σημάνει κάτι μια τέτοια εξέλιξη στις κοινωνίες μας. Ωστόσο, ε, παρόλο που δεν, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τα πάντα από τώρα, είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσουμε ορισμένα δύσκολα θέματα ή και προβλήματα. Κοινωνικός διάλογος δίνεται πολύ μικρή ε, προσοχή ε, σε αυτό το θέμα. Κάποιοι κοινωνικοί εταίροι έχουν δραστηριοποιηθεί και όπως συμβαίνει συνήθως στη βιομηχανική πολιτική, ε, αυτό αντικατοπτρίζεται και στο σύστημα των μαθητιών. Ωστόσο, η μόνη χώρα στην οποία κάτι κινείται είναι η Γερμανία, όπου υπάρχει και η πρωτοβουλία βιομηχανία 4.0. Οι νέες εταιρείες έχουν συνήθως λιγότερους αλλά πιο καταρτισμένους εργαζόμενους και αυτό αποτελεί πρόκληση για τον κοινωνικό διάλογο και το μέλλον του κοινωνικού διάλογου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να διεξαχθεί κοινωνικός διάλογος σε αυτόν τον τομέα. Αντιθέτως υπάρχουν πολλοί εκπρόσωποι και από κράτη-μέλη ε, όπου υπάρχουν ε, οργανωμένοι ε, κοινωνικοί εταίροι και όπου ο κοινωνικός διάλογος λειτουργεί κανονικά και αποτελεσματικά. Έχουμε και άλλο ένα έργο για την επιχειρηματικότητα και τις μικρομεσίες επιχειρήσεις και τη διεθνοποίησή τους. Ε, στιάζεται στις εκφύσεως παγκοσμιοποιημένες επιχειρήσεις που από, από την αρχή της ύπαρξής τους έχουν εμπλακεί σε διεθνείς δραστηριότητες. Είναι νέες, νεοφύης επιχειρήσεις, καινοτόμες και διεθνείς παγκοσμιοποιημένες δηλαδή ε, δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον δύο χώρες με όσον αφορά τι πωλήσει του και τον κύκλο εργασιών του. Και αυτό που θέλουμε να ερευνήσουμε με αυτό το έργο είναι αφενό ποιο είναι ο ρόλο του στι ε, παγκοσμίε ε, αλυσίδε προμηθειών ε, και πώ σχετίζονται με την δημόσια πολιτική. Και αυτό που βρήκαμε εδώ για αυτές τις Born Global το, στο επιχειρηματικό τους μοντέλο η διεθνοποίηση είναι κλειδί, είναι μια κομμάτι του επιχειρηματικού του σχεδίου οι λειτουργικές τους ε, πτυχές εστιάζονται στις διεθνεί ε, συναλλαγές κυρίως διότι εμπλέκονται στην ανάπτυξη ειδικευμένων καινοτόμων προϊόντων για τα οποία η εθνική αγορά, η εγχώρια αγορά θα ήταν πολύ μικρή, οπότε για να είναι βιώσιμες και ανταγωνιστικές πρέπει να διεθνοποιηθούν. Είναι αρκετά μικρές. Στις επιχειρήσεις που μελετήσαμε εμείς ε, έχουμε μεταξύ 5 και 110 επαλλήλων, αλλά είναι πολύ δυναμικές όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασία. Επίσης οι συνθήκες εργασίας φαίνεται να είναι αρκετά καλές ε, σε αυτές τις επιχειρήσεις. Το ίδιο και η ποιότητα του εργατικού δυναμικού υψηλά καταρτισμένο και εκπαιδευμένο και νέοι σε ηλικία. Έχουν διαφορετικές θέσεις ε, στην αλυσίδα ε, προσφοράς και αξίας, αλλά διευκολύνουν και άλλες επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στην αλυσίδα παραγωγής, στην αλυσίδα παροχής όσοι συνεργάζονται με αυτές ε, αποκομίζουν αμοιβαία ωφέλη. Αλλά αυτά τα αμοιβαία ωφέλη εξαρτώνται από τις αλυσίδε ε, και τους υπόλοιπου συμμετέχοντες, τις, ποιες είναι οι σχέσεις τους ε, μεταξύ των εταιρείων αυτών. Όσον αφορά αυτές τις εκφύσεως παγκόσμιες επιχειρήσεις, είναι πιο ανταγωνιστικές, πιο βιώσιμες έχουν βελτιωμένη πρόσβαση στις αγορές και σε δίκτυα. Οι αλυσίδε ε, προμηθείων επίση βοηθούν να βελτιώνουν τα προϊόντα και τις διαδικασίες τους. Έχουν λοιπόν μακροχρόνιες προοπτικές. Όσον αφορά τις πολιτικές, αυτό παρατηρούμε γενικότερα είναι μια μεγάλη ποικιλία υποστήριξης της διεθνοποίησης ε, στην Ευρώπη, τόσο από κυβερνήσεις, κοινωνικούς ατόερου, δηλαδή δημόσιους φορείς, που μέσω πολιτικών και στρατηγικών ε, ε, ε, ε, διαθέτουν σε επιχειρήσεις διάφορα μέσα υποστήριξης εστιάζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως αλλά αυτή η συγκεκριμένη ομάδα των μικρών διεθνών νεοφιών επιχειρήσεων είναι κάτι ιδιαίτερο. Έχουν πιο συγκεκριμένες ανάγκες, οπότε μπορεί να υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Επίσης, αυτό που ακούμε από την ανάλυση πολιτικής είναι ότι μέτρα υποστήριξης διεθνοποίησης ε, όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στη δικτύωση ε, χρειάζεται ιδιαίτερη προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η παρακολούθηση επίσης και η αξιολόγηση είναι πάρα πολύ σημαντική από αυτή την άποψη. Ένα άλλο πρόβλημα παρατηρούμε είναι ότι παρότι υπάρχουν όλα αυτά τα μέσα διαθέσιμα, πολλέ επιχειρήσει δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει διαθέσιμο για αυτές στην αγορά. Δεν φαίνεται να προωθούνται, να προβάλλονται παρκώ ε, τα εργαλεία στι εταιρείε, ούτε να του είναι απόλυτα κατανοητά. Δεδομένου ότι έχουν και πολλέ διαφορε μεταξύ του, οπότε είναι δύσκολο να καταλάβουν ποιο από τα διαθέσιμα μέσα τη συμφέρει περισσότερο μια άλλη πτυχή αρκετά γνωστή, ο διοικητικός φόρτος εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για τις μικρές επιχειρήσεις παρόλε τις δραστηριότητες των τελευταίων ετών. Αλλά ακόμη και με όλα σε αυτά τα μέσα στήριξης φαίνεται να εξακολουθεί να είναι πρόβλημα ο διοικητικός φόρτος. Ε, πρόβλημα και για τις επιχειρήσεις και για τους διαχειριστές αυτών των μέσων. Έχουμε Ξε, ξεπεράσαμε λίγο τα όρια, οπότε κάπου εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ πολύ να ευχαριστήσω τον κύριο Στόρι και την κυρία Μάντελ. Και τώρα θα δώσω το λόγο για ερωτήσεις, παρεμβάσεις από τα μέλη μας εδώ. Ενδεχομένω και τους συντονιστές. Δεν είναι εδώ συντονιστής βέβαια για ζητήματα απασχόληση του ΕΛΚ. Είναι όμως εδώ η Άγνες Γιονκύρης ε, από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Μπορείτε να θέσετε ένα ερώτημα παρακαλώ. Σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό ερώτηση. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστώ πάντως πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ευχαριστώ και για αυτό το έτσι τόμο με πληροφορίες. Ε, δεν μπορούσα να το διαβάσω ακόμα. Ε, έχω τρία σύντομα ερωτήματα και ελπίζω να μπορέσετε να με διαφωτίσετε. Πρώτον, θα ήθελα να μιλήσουμε για το θέμα της συμμετοχής των εργαζομένων ε, στις, στο εταιρικό δίκαιο με βάση τις νέες τεχνολογικές μορφές βλέπουμε ότι είναι όλο και πιο εξατομικευμένες οι θέσεις ε, ε, οι σχέσεις μάλλον εργασίας. Ε, μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο για την εκπροσώπηση των εργαζομένων σε αυτές τις νέες θέσεις απασχόλησης. Δεύτερον, στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται ε, κάποια στοιχεία ποιοτικά για τις θέσεις απασχόλησης Δηλαδή τι είδου θέσει εργασία αυτέ που επανέρχονται στον τομέα τη μετοποίηση, διότι καλό είναι να επιστρέφουν οι θέσει εργασία στην Ευρώπη, αλλά να μην οργανώσουμε έτσι μια κούρσα προς τα κάτω και μια ισοπαίδωση. Και το τρίτο θέμα είναι το θέμα της εκπαίδευσης. Αυτό σχετίζεται και με την περιφερειακή πολιτική κατά κάποιο τρόπο. Διότι αν δούμε πώς είναι η κατάσταση στην Ευρώπη, κάποιες περιφέρειες έχουν πληγεί πολύ περισσότερο από την αποβιομηχανοποίηση ε, και συχνά οι ίδιες αυτές περιφέρειες ε, είναι αυτές που δεν έχουν και οικονομικά μέσα. Ακριβώς δηλαδή στις περιοχές εκείνες ε, όπου πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση, κατάρτιση, μάθηση ε, για τους εργαζόμενους. Ε, ε, πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα και, το, και επίσης και το κενό, η απόκληση που υπάρχει μεταξύ της, των δεξιοτήτων και των θέσεων απασχόλησης. Εάν μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια από αυτών των ζητημάτων, θα ήμουν ευγνώμων. Μάλιστα, θα έχουν δύο λεπτά και οι υπόλοιποι η κυρία Μάκιντάιρ από το ECR στις τρία θέματα Πασχόλησης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της επιστροφής των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Έγινε και μια ακρόαση του Σεπτέμβριο του 2015 από την Επιτροπή Απασχόλησης ε, για αυτό το θέμα. και τότε ασχοληθήκαμε με τους επιμέρους παράγοντες, ε, την σημασία της ε, μείωσης του ενεργειακού κόστους. Ε, ήταν κάτι που είχε τονιστεί ιδιαίτερα αυτό. Όπως ήδη ελέγχθη το θέμα των δεξιοτήτων και η έλλειψη συγκεκριμένων δεξιοτήτων, βασικών δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Επίση, ο συσχετισμός μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων και η σημασία του να μειωθεί, η ανάγκη μάλλον, μάλλον να μειωθεί το διοικητικό άξονα το ρυθμιστικό άχθος τη μικρομεσαία επιχείρηση. Δηλαδή ε, προσπαθούμε να απλοποιήσουμε ε, την νομοθεσία. Αυτός είναι ο σκοπός. Όχι να μειώσουμε την προστασία των εργαζομένων, αλλά πρέπει να απλοποιήσουμε του νόμου, Δηλαδή μια μικρή επιχείρηση να μην πρέπει ε, να επιβαρύνεται με δικηγόρους, ε, με διάφορους ε, μεσάζοντες. Γίνεται συχνά λόγος για καλύτερη νομοθεσία προς την κατεύθυνση αυτή. Ό,τι αφορά τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης που επέστρεψαν ε, λένε, λέμε εμείς στη Βρετανία ότι προσέχουμε τα cents, μετά τα ευρώ, προσέχουν τον εαυτό τους. είναι λίρες το λέμε αυτό βέβαια. Ε, μόνο το Μάρτιο φέτος ε, η Vodafone επέστρεψε 2.100 θέσεις εργασίες. Ε, σιγά σιγά λοιπόν υπάρχει μια επιστροφή. Οι περισσότερες εταιρείες οι οποίες ακολουθούν αυτή τη διαδικασία θεωρούν ότι τα βασικά στοιχεία που το οποία τους κάνουν αυτό είναι η ποιότητα αλλά και η εγκύτητα. Είναι πολύ πιο εύκολο ε, να πάρει κανείς τηλέφωνο κάποιον που μένει απέναντι για να ζητήσει να του παραδώσουν κάτι από ότι να στείλει ένα mail στην Κίνα και να περιμένει κάποιε εβδομάδες. Δηλαδή είναι σημαντικό να μειωθεί και η αλυσίδα διανομής και στον Ηνωμένο Βασίλειο ε, η οργάνωση των μεταποιητών λένε ότι υπάρχουν και κάποιες ανησυχίες ε, σε ό,τι αφορά την ποιότητα και γι' αυτό υπάρχει η επιστροφή ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις ε, ε, πολλές λένε ότι η, ποιότητα είναι ο βασικός παράγοντας για την επιστροφή τους. Έτσι λοιπόν το, το περιβάλλον που δημιουργούμε εμείς στην Ευρώπη θα πώς μπορεί να βοηθήσει τη μεταποίηση να στεφθεί από επιτυχία στην παγκόσμια οικονομία. Ω πολιτικοί ηθήνοντες ποια μέτρα πιστεύετε ότι μπορούμε εμείς και πρέπει να θεσπίσουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα περιβάλλον το οποίο θα βοηθήσει τη μεταποίηση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η κυρία Βίμη, που είναι μέλος και των δύο επιτροπών, έχει εδώ λόγο. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του κυρίου Καλβέτζαμπο. Δύο θέματα. Ποιος είναι ο αντίκτυπος, αν υπάρχουν, αν υπάρχει τέτοιος, από την Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση, ιδίως του ΕΤΣΕ, στη διάρκεια της ε, μελέτης τους βλέπουν ότι υπάρχει σκοπευμένη χρήση του ΕΦΣΙ και άλλων χρηματοδοτικών μέσων για να υποστηριχθούν τομεί όπως η ψηφιοποίηση των μικρονομικών επιχειρήσεων, η ανθεκτικότητά τους στην ε, παγκοσμιοποίηση και ποιοι τομείς μπορούν να συμβάλλουν ε, στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Επίσης, η μεταποίηση και οι υπηρεσίες ε, αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια ε, σημαντικά. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τη δική σας παρουσίαση για τις τεχνολογίες που αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού, του παιχνιδιού τα επόμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι θα, ότι θα απαιτηθούν νέοι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι ε, με ε, πανεπιστημιακά πτυχία, αλλά και ότι οι εργάτες θα χρειάζεται να επανακαταρτίζονται προκειμένου να ε, διατηρηθεί ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα της μεταποίησης. Μπορείτε να μας περιγράψετε ποιοι τομείς ε, στον, στον κλάδο της μεταποίησης παρουσιάζουν το μεγαλύτερο δυναμικό, δυναμικό για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πιστεύετε ότι οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να συνεργαστούν προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσει αυτών των νέων τεχνολογικών εκκλήσεων και έχετε ε, παραδείγματα των πρακτικών που ήδη βρίσκονται στο στάδιο της εφαρμογής. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα επανέλθουμε στους εμπειρογνώμονές μας και θα τους ζητήσουμε να απαντήσουν ε, στις ερωτήσεις. Ναι, ήταν πολύ καλές οι ερωτήσεις. εγώ ως ε, αρχαιότερος θα απαντήσω στις εύκολες ερωτήσεις και θα αφήσω τους συναδέλφους τις δύσκολες. Λοιπόν, για την συμμετοχή των εργαζομένων. Δυστυχώς ε, φαίνεται ότι είναι δύσκολο το θέμα αυτό στον τομέα της μεταποίησης. Ωστόσο, οι νεοφυείς επιχειρήσεις, σε όποιον κλάδο και αν το δούμε, ε, δεν, πολύ συχνά ε, δεν συνειδητοποιούν ε, στα πρώτα στάδια το, της δραστηριότητάς τους την ε, αξία και τη σημασία της συμμετοχής των εργαζομένων. Ωστόσο, εγώ θα ανησυχούσα πιο πολύ για την συμμετοχή των εργαζομένων όσον αφορά τις διαρθρωτικές, τις δομικές αλλαγές που επίκυνται Γι' αυτό και χρειάζεται καλύτερη πληροφόρηση, καλύτερη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων, διότι αυτά τα θέματα είναι θέματα που θα επανέρχονται τις επόμενες δεκαετίες, δηλαδή συμμετοχή εργαζομένων ε, και συμμετοχή του στη λήψη αποφάσεων είναι αναγκαία και απαραίτητη ε, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης ε, της, του κλάδου της μεταποίησης. Ποιότητα των θέσεων εργασίας που επιστρέφουν. Κυρία Μάκιντάιρ, επιβεβαιώνω αυτό που λέτε κι εσείς. Το κίνητρο για την επανεγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη είναι η εγκύτητα βεβαίως, αλλά ε, πολύ συχνά ε, έχουμε διαπιστώσει ότι είναι και η διασφάλιση της ποιότητας. Αυτές οι απομακρυσμένες δραστηριότητες, όπως είναι τα call center για παράδειγμα, ε, έδειξαν ότι πολλές φορές δεν μπορούσε να διασφαλιστεί η ποιότητα. Και αυτός είναι μακράν ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο επιστρέφουν πολλές δραστηριότητε στην Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες λοιπόν ε, ξέρουν και εκτιμούν ε, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των Ευρωπαίων εργαζομένων, γι' αυτό και αμείβονται ε, αξιοπρεπώς οι θέσεις εργασίας αυτές. Και να πω επίσης ότι ίσως διέτρεξα πολύ γρήγορα τις ε, διαφάνειες, αλλά ε, πράγματι και με βάση τις δικές μας έρευνες ε, η περίπτωση της Vodafone είναι το, το, το, το καλύτερο και το μεγαλύτερο παράδειγμα επιστροφής. Ποιες είναι οι πολιτικές που πρέπει να ακολουθήσουμε τώρα. Είμαστε λίγο επιφυλακτικοί στο να δώσουμε συγκεκριμένε συστάσει ω προ το ποιε θα πρέπει να είναι οι πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθούν. Συνήθως εμείς μιλούμε για επιλογές πολιτικής. Ε, δίνουμε ορισμένες ε, κατευθυντήρες γραμμές δηλαδή. Δεν θα ήθελα να είμαι πολύ συγκεκριμένο. Ωστόσο, για το συγκεκριμένο ζήτημα της επαναγκατάστασης βιομηχανικών δραστηριοτήτων, θεωρώ ότι αν είναι να καταρτιστεί μια συγκεκριμένη στρατηγική βιομηχανική, θα πρέπει να υπάρξει και ένας έλεγχος. Όπως είπα και εισηγητικά, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία δεν έχουν μια συγκεκριμένη τέτοια πολιτική ελέγχου. Αν λοιπόν πραγματικά ε, θέλεις να, να επαναφέρεις βιομηχανικές δραστηριότητες στην Ευρώπη πρέπει να καταρτήσεις και συγκεκριμένη πολιτική για το πώς θα φτάσεις σε αυτόν τον στόχο και να στελεχώσεις τις αντίστοιχες υπηρεσίες με επαρκές προσωπικό. Αυτά από μένα. Εγώ θα απαντήσω στις άλλες ερωτήσεις, αλλά θέλω να πω κάτι όσον αφορά την εκπροσώπηση των εργαζομένων. Αυτό που βλέπουμε με τις ε, νεοφυείς επιχειρήσεις ε, διεθνούς χαρακτήρα, βλέπουμε ότι τελικά η εκπροσώπηση δεν είναι τόσο μεγάλο ζήτημα, διότι εμπλέκονται άμεσα, συμμετέχουν άμεσα εργαζόμενοι. Θεωρούνται όχι απλά ως ε, εργαζόμενοι, Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη μετάφραση το οποίο επιλύθηκε λοιπόν. Οπότε τελικά δεν απαιτείται να υπάρχει κάποιο σωματιο εργαζομένων διότι υπάρχει άμεση συμμετοχή των εργαζομένων κάτι που είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους νέους ανθρώπους αυτού του νέου τύπου εταιρείες. Συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Από την άλλη, αυτό που παρατηρούμε όσον αφορά τις ρεξικέλευθες τεχνολογίες, την ψηφιοποίηση, πριν από δύο χρόνια η Eurofund έκανε ένα άλλο έργο που ονομαζόταν νέε μορφές εργασίας». Εκεί συζητήσαμε για διάφορους νέους τύπους οργάνωσης των εργασιών και σχέσεις ε, ε, εργαζομένων είδαμε ότι όλα αυτά επηρεάζουν θετικά την εκπροσώπηση των εργαζομένων. Είναι τόσο νέε αυτέ οι μορφέ που δεν καλύπτονται τι παραδοσιακέ. Με στα επόμενα δύο χρόνια λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιε θα είναι οι εξελίξει, ποιε νέε ε, δομέ διαλόγου θα δημιουργηθούν. Όσον αφορά την κατάρτιση και την εκπαίδευση, αυτό που βλέπουμε στις περιοχές που εμείς αναλύσαμε στο πρόγραμμά μας, στο έργο μας, είναι ότι οι περισσότερες περιφέρειες, περιοχές δεν έχουν εντολή για να θεσπίσουν πολιτικές εκπαιδευτικές είτε από εθνικό είτε από περιφερειακό επίπεδο. Το μόνο παρατηρούμε, που παρατηρούμε εκεί είναι ότι όσον αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ε, εκπαίδευση η περιφερειακή πολιτική συνδέεται έμεσα. Αλλά υπάρχουν άλλα παραδείγματα όπου οι περιφερειακοί παράγοντες κατάφεραν να επηρεάσουν επιτυχώς τα προγράμματα σπουδών πανεπιστημίων ε, ή κέντρων ε, επαγγελματικής κατάρτισης. Ιδανικά αυτό θα έχει συνέπειες και στο εθνικό επίπεδο, οπότε είναι αμφίδρομη η ανταλλαγή. Όσον αφορά το κανονιστικό φόρτο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σίγουρα έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος την τελευταία δεκαετία. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ακόμη, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι τελικά πράγματα που είναι χρονοβόρα για μικρομεσαίες και για μεγάλες επιχειρήσεις είναι επίσης χρονοβόρα για τις μικρές επιχειρήσεις λόγω περιορισμένων πόρων και λόγω τη έλλειψη ειδικευμένων ε, τμήματων σε μικρέ επιχείρησει που να μπορούν να ασχοληθούν ειδικά με αυτά τα ζητήματα. Οπότε και εκεί υπάρχουν ζητήματα προ αντιμετώπιση. Αυτό παρατηρούμε εδώ όσον αφορά τα μέσα υποστήριξη τη παγκοσμιοποίηση και τη διεθνοποίηση είναι ότι οι online διαδικασίε ε, φαίνεται να βοηθούν και τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, όταν μπορούν να συμπληρώσουν κάποιο έντυπο online αυτό τους γλιτώνει χρόνο μπορούν να το εντάξουν εύκολα στις κανονικές διαδικασίες τους. Όσον αφορά και την ομοθεσία, εκεί τίθε το ζήτημα του περιβάλλοντος πολιτικής. Κάτι άλλο σημαντικό είναι η σταθερότητα ώστε οι επιχειρήσεις να μην έχουν να κάνουν διαρκώς με νέες εξελίξεις και νέες αλλαγές στις οποίες πρέπει να προσαρμοστούν. Όσον αφορά την επίδραση των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων και Επενδύσεων, Υπάρχουν κάποια καλά παραδείγματα όπου ο ρόλος τους ήταν κλειδί στην περιφερειακή πολιτική, κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε περιοχές Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ περιφερειών, την ανταλλαγή εμπειριών, διδάγματα που βοηθούν. Και επίσης έχουμε κάποια παραδείγματα συνεργασίας κοινωνικών εταίρων και στα δύο έργα για τα οποία μίλησα, για την περιφερειακή πολιτική αλλά και για την υποστήριξη προς τη διεθνοποίηση, παρατηρήσαμε ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά αν δεν προέρχονται μόνο από κυβερνήσεις αλλά από τριμερείς οργανισμούς, ένα συντονισμένο, συντονιστικό οργανισμό ε, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους κοινωνικούς εταίρους. Είναι προφανές για όλους μας ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα και ήμασταν πολύ αποτελεσματικοί. Έχουμε ακόμα 7 λεπτά για αυτήν τη συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Σίμπεν Τόμας, ο οποίος είναι ε, υποδιευθυντής ε, της σχετικής μονάδας. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν περίμενα να μου δώσετε το λόγο. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Πάντως, ε, ε, για το θέμα που, που αναφέρθηκε η χρηματοδότηση και στα πλαίσια του ΕΦΣΥ υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή εκεί υπάρχει άλλη μια πηγή χρηματοδότησης. Ε, θα ολοκληρωθεί στον επόμενο 1,5 έτος αυτό το πρόγραμμα. Όπως είπαν οι συνάδελφοι στο πάνελ υπάρχουν ακόμα κάποια ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, ε, η ανάπτυξη ε, των διαφόρων σεναρίων για την απασχόληση των ε, ε, το θέμα των μισθών και της παραγωγικότητας ε, θα αναφέρονται εκεί, αλλά και κάποια ακόμα περιφερειακά σεμινάρια που θα λάβουν χώρα, μεταξύ των οποίων σεμινάρια που θα διαδώσουν τα ευρήματα σε ό,τι αφορά ε, τις διάφορες πολιτικές επιλογές αναομάδες χωρών της Ένωσης θα γίνουν αυτά τα σεμινάρια. Επίσης υπάρχει και μια έμεση διασύνδεση με την κοινο, και, ανακοίνωση ε, για την πολιτική βιο, τη βιομηχανική. Ε, ελπίζουμε και αυτό να έρθει να τροφοδοτήσει αυτές τις δράσεις, τα προφίλ των δεξιοτήτων ε, και άλλα σχετικά ζητήματα. Αναμένουμε με ανυπομονησία της νησφοράς σας για να μπορέσουν αυτά τα project να τελεσφορήσουν. Ευχαριστώ. Okay. Uh, Ωραία. Συγγνώμη που ε, κάποιοι μόλις καταφέρατε να φτάσετε. Ξέρω ότι είναι Δευτέρα και ότι υπάρχουν προβλήματα ε, στο να φτάσει κανείς έγκαιρα. Έχουμε πολύ λίγα λεπτά όμως που μας απομένουν. Ποιος θέλει το λόγο για να κάνει μια τελευταία παρατήρηση, παρέμβαση σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ε, Mr. Ε, Κύριος Μαρτάν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, φοβήθηκα ότι δεν θα έπαιρνα το λόγο τελικά. Άκουσα πολύ προσεκτικά τους εμπειρογνώμονες της Eurofound και θέλω να τους ευχαριστήσω για τη μελέτη τους και για την παρουσίασή τους. Όμως ε, δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι το Eurofound εδώ απαντά σε μια παραγγελία, σε ένα αίτημα της Κομισιόν. Και η Κομισιόν, όπως ξέρουμε, έχει μεγάλο πόνο με την ε, ένταξη της Ευρώπης στην παγκοσμιοποίηση και στην παγκόσμια αγορά και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Και πρέπει εμείς να συνοδεύσουμε αυτή την παγκοσμιοποίηση. Πρέπει να μην χάσουμε το τρένο, αλλιώς θα τα χάσουμε όλα. Αυτό μας λένε. Και εδώ είναι που δεν συμφωνώ καθόλου μαζί σας, ε, κύριε εμπειρογνώμονες. Δηλαδή, εσείς, το, όλος τρόπος σκέψης σας εγγράφεται σε αυτό το πλαίσιο. Η παγκοσμιοποίηση όμως τι είναι. Φτιάχνουν σκλάβοι στον τρίτο κόσμο προϊόντα και τα πουλούν στους άνεργους στην Ευρώπη. Αυτό είναι. Ε, ε και οι μικρομέσες επιχειρήσεις μας ενοχλούν. Καλύτερα να βοηθήσουμε τη startup που ήδη έχουν σκεφτεί να, ότι πρέπει να, εργαστούν διεθνώ. Μην ξεχνάτε όμω ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οι μικρέ επιχειρήσει εκπροσωπούν 90% των θέσεων απασχόληση, των μισθωτών θέσεων απασχόληση. Αν χάθηκαν 3 εκατομμύρια, εκατομμύρια θέσει εργασία από το πρώτο που ξεκίνησε η κρίση, αυτό έχει να κάνει με το δόγμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για έναν ελεύθερο και ε, χωρί εμπόδιο ανταγωνισμό. Τι θα γίνει, πώ θα προστατεύσουμε όμω τι μικρομεσαίε επιχειρήσει μα που εκπροσωπούν να παραλαμβάνουν 90% των θέσεων απασχόληση, γιατί να μην προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τις δικές, τη δική μα εσωτερική αγορά που υπάρχει απέναντι στον τον ανταγωνισμό, τον αθέμητο ανταγωνισμό από όλο τον κόσμο. Ε, αυτά είναι τα ερωτήματα που είχα να θέσω, που θα ήθελα να σα είχα θέσει μάλλον, γιατί είναι μάλλον αργά. Ε, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλε ερωτήσει, κύριε Μαχτά. Δεν ξέρω πότε γεννηθήκατε, αλλά εγώ γεννήθηκα στην καρδιά του 50 και εσείς ε, δίνετε επιχειρήματα, αλλά και γεννήθηκατε και εσείς στην καρδιά του 50. Ε, είναι τελείως διαφορετική εποχή όμως τότε. Δεν μπορείτε να λέτε πια θα καταπολεμήσω την παγκοσμιοποίηση. Οι τεχνολογικές, οι οικονομικές αλλαγές δεν μπορούμε να πολεμήσουμε. Πρέπει όμως να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε να είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι οι πολίτες, ε, να έχουν ισχύ στον τόπο, τρόπο, τον τόπο εργασίας τους, στον χώρο εργασίας τους, ε, με δικαιώματα και με ισότητα. Για μια καλή ε, εργασιακή ζωή με καλά οικονομικά αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στα 150 και γι' αυτό έγινε και αυτό το σεμινάριο. θα, σίγουρα θα πρέπει να ξαναγίνει και άλλο τέτοιο σεμινάριο. Βέβαια, το επόμενο βήμα είναι το τι θα κάνουμε επακριβώς τώρα για να διαφυλάξουμε την αγορά εργασίας όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και εκτός Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή την σύντομο, το σύντομο αλλά ε, έτσι ε, ιδιαίτερα ζωηρό σεμινάριο.